πρώτη έκθεση είναι του κυρίου Φερέιρα. Ο εισηγητής έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πριν από την ψηφοφορία να υπογραμμίσω ότι η πολιτική μας ομάδα είχε προτείνει γενικά μια συζήτηση για την αλληλεία γενικότερα που θα συμπεριλαμβάνει και το θέμα της συμφωνίας της αλλιευτικής με το Σάουτο Μέι Πρίντσιπε. Αλλά οι μεγάλες πολιτικές ομάδες, οι περισσότερες μάλλον πολιτικές ομάδες αρνήθηκαν να γίνει μια τέτοια συζήτηση. Αν και δεν είχαμε ιδιαίτερα βεβαρημένη θα έλεγα ημερήσια διάταξη, είχαμε και πολλά κενά θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, βασικό στόχος είναι να δούμε εδώ πώς θα μπορέσει το Κοινοβούλιο να ξεπεράσει αυτόν τον ρόλο τον άχαρο που έχει, που μπορεί να πει ή ναι ή όχι μόνο στην συγκεκριμένη πρόταση. Θα έπρεπε να μπορέσουμε να κάνουμε μία συζήτηση επί της ουσίας. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μία σωστή τροποποίηση της φιλοσοφίας και των στόχων της συγκεκριμένης συμφωνίας. Έχει σημασία λοιπόν να εγκρίνουμε την πρόταση και για το ΣΑΟΤΟΜΕΙ Μέι πρίνσιπε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για να καλύψουμε αν θέλετε το, τον αρνητικό απολογισμό της προηγούμενης συμφωνίας. Πρέπει να βελτιώσουμε φυσικά την αξιοπιστία των στατιστικών και των αριθμών για τα αλλιεύματα, θα πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα τα διαθέσιμα αλλιεύματα, και να βοηθήσουμε την άλλη πλευρά. Να υπάρξει σωστή συνεργασία, ξεπερνώντας όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, οι οποίες μας έχουν ε, οδηγήσει σε μια ουσιαστική απόκληση ε, από τις βασικές αρχές ε, μιας διμερούς συμφωνίας. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια σωστή αλλαγή για τη χώρα αυτή και για μας. Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Περνάμε τώρα σε ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται η ψηφοφορία. Has everyone voted? Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκτή η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η επόμενη έκθεση, Καντέκ, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες; Δεκτή η πρόταση. Συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Μπροκ. Και εδώ ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίες; Δεκτή η πρόταση. Περνάμε τώρα στη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή για τις μεταφορές και τον τουρισμό. Μία ψήφος για Ανατάσσεως χειρών. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή η πρόταση, μαζικά ευχαριστώ. Η επόμενη ψηφοφορία είναι η έκθεση της κυρίας Ρης, η τελευταία συζήτηση που κάναμε για τα γενετικά τροποποιημένα. Θα ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση για την τροπολογία 52. Σας θυμίζω ότι απαιτείται ειδική πλειοψηφία εδώ, 356 ψήφων. Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 52. Πέρα στη ψηφοφορία, συνάδελφοι. And that has been adopted by... 480 υπέρ. Υπάρχει ειδική πλειοψηφία. Λοιπόν, έχει τροποποιηθεί η θέση του Συμβουλίου. Η επόμενη ψηφοφορία είναι η έκθεση ΜΑΤΟ για την αλληλεία και αυτή. Θα ψηφίσουμε τώρα τις τροπολογίες 1 με 2 και 4 με 25. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Δεκτές. Τώρα, τροπολογία 26. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 28. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθεται. Ψηφίζουμε για την πρόταση της Επιτροπής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τώρα, ονομαστική κλίση για το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας, δεκτή η πρόταση. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες για σήμερα και τώρα θα ξεκινήσουν οι επεξηγήσεις.